Παρακαλώ καθίστε και ετοιμαστείτε για την ψηφορία. Η πρώτη ψηφορία. Αφορά την έκθεση Σικιαρχική. Για το ποσοστό αναπροσαρμογής για άμεσες ενισχύσεις. Για το 2015. Μία και μόνη ψηφορία και ονομαστική. Ψηφίζουμε. Where see? maybe allow people to arrive a bit. I give people 30 seconds to arrive. Σας δίνω μισό λεπτό για να καθίσετε και να ψηφίσετε παρακαλώ. So, now I can do this, system. Yeah, still. When we get to what, 700? get to 700? Mr. Brooks. Come on. I think we can. Okay. Yeah. Okay. The vote is closed. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η επόμενη ψηφοφορία σημαίνει όσον αφορά την στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σώτα ανδρών γυναικών μετά το 2015. Η πρώτη ψηφοφορία είναι ένα εναλλακτικό ψήφισμα με ανάταση χειρών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψήφισμα. And the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτωται. Now, colleagues, we now come to the split votes and we come to paragraph 1. Τώρα με τις χωριστές ψηφοφορίες, πρώτη παράγραφος, το αρχικό κείμενο σε δύο ψηφοφορίες, το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη παράγραφο Σε δύο τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Νομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας και αυτή εγκρίνεται. Παραγραφός 5, δύο τμήματα. Πρώτο, ανάταση χειρός. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίνεται. Παράγραφος 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Έλεγχος για το 8. Ψηφίζουμε. σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκλίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκλίνεται. Παράγραφος 11. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκλίνεται Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Σε τρία τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 28. Σύνδεο τμήματα το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Τρία τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος ψηφίζουμε Πέρασε. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα. Τρία τμήματα το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίση. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρα. Εγκρίνεται. 41. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 τέσσερα τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το τρίτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Μια ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Τρία τμήματα το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτωται. Έλεγχος για το 59 τρίτο τμήμα. Ψήφιζουν. πέρας απορρίπτεται καθαρή διαφορά παράγραφος 60 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. 67. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Οκτώ. Σε τέσσερα τμήματα το πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 72. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για το 73 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 του μετά το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και λογικές ε, διατάξεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 18 τώρα παράγραφος 30 υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται παράγραφος G αγγλικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος L σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης εν νι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος όμικρον σε δύο τμήματα υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική π. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Επαληθεύουμε. Αιτιολογική π, δεύτερο τμήμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Αιτιολογική S, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, τρία τμήματα, συγγνώμη, κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Αιτιολογική v Υπέρ κατά αποχές. Επίσης εγκρίνεται ψήφισμα στο σύνολό του, ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. And the vote is closed. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια κυρία Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια και συνεχίζουμε. Δύο εκθέσει ακόμα. Η πρώτη τη κυρία Μόσκα, δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία σε τρίτε χώρε πρώτη παράγραφους 5, υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 13, δύο τμήματα, πρώτο υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται Επίση, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται επίσης 37 ε, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 40 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται παράγραφο 42 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. αντιλογική σκέψη 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται. Ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. και εγκρίνεται. Και τώρα τελευταία έκθεση, έκθεση Σφόμποντα. Δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρώτη παραγωγή 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχέ. Επίση. 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 σε δύο τμήματα. Υπέρ για το πρώτο. Δεύτερο, κατά. Αποχές. Δεύτερο, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία για το ψήφισμα στο σύνολό του. Ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα διακόπτουμε αγαπητοί συνάδελφοι έως τις 12 και 30, αλλά παρακαλώ να παραμείνετε στην αίθουσα για την πανηγυρική συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Μογγολίας. Okay. <laughs> I'll take my coffee with me.